May I ask all the people who are standing up to just have their seats. Παρακαλώ να καθίσετε για να αρχίσει η ψηφοφορία. Down. Keep quiet because we are going to start. Παρακαλώ καθίστε για να αρχίσουμε. Okay. As uh, it Όπως είπαμε και χθες και συμφωνήσαμε, θα αλλάξουμε ε, και την σειρά με την οποία θα ψηφίσουμε κάποια θέματα. Αρχίζουμε το 15 και 16 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ο εισηγητής κύριος Τζανλούκα Σούστα ζήτησε το λόγο. Τζανλούκα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, θα ήθελα να σας ζητήσω κατά πόσο θα ήταν δυνατόν να έχουμε split votes στις προφορικές τροπολογίες που θα παρουσιάσει ο συνάδελφος Άνσλικ. Μιλάμε για 79-64. Ε, σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις και τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας, η θετική ψήφος που έχει συμπεριληφθεί στην λίστα ψηφοφοριών θα πρέπει να αναφέρεται στο αρχικό κείμενο. Μιλάμε για τι τροπολογίε 79 και 64 στου δύο φακέλους και όχι για τη νέα προφορική τροπολογία. Και, στην... και να μην αναφέρεται στη νέα προφορική τροπολογία. Ευχαριστώ. Πολύ καλά, το σημειώνω. Και όταν φτάσουμε στη προφορική τροπολογία θα επανέλθουμε. Δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Προφορικές Τροπολογίες. Λοιπόν, σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Γνωμοδότηση για την ΙΜΚΟ πρόκειται για νομοθετικού περιεχομένου γνωμοδότηση. Επί της ουσίας, υπεύθυνη είναι η ΙΜΚΟ. Το θέμα μας, όπως ξέρετε, αφορά πρόταση για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση τη 42. Αρχίζει η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση Τις 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι. Παρακαλώ. Μόνο τα μέλη της Επιτροπής δικαιούνται να ζητήσουν ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ηλεκτρονική επαλήθευση της 54. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 55 και 56 on block. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 58, 59, 60 και 61 on block. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονική επαλήθευση κάνουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Έχουμε κάποιον από την ECR Να ψηφίζουν ε, παρακαλώ οι ίδιοι κάθε φορά για να μην δυσκολευόμαστε. Λοιπόν, έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 65. Αρχίζει ψηφοφορία. ένας παραπανήσιος σοσιαλιστής. Παρακαλώ. Εντάξει. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση 66. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 68. Εγκρίνεται. Πρώτη συμβαστική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εβδομήντα οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79. Έχουμε την ε, προφορική τροπολογία της κυρίας Δεσαρνέζ. Υπάρχει αντίρρηση? Έχετε στο φάκελό σας το κείμενο. Ζητήθηκε από τον Τζανλούκα Χωριστή ψηφοφορία. Την 79. Έχετε την ε, διατύπωση της προφορικής τροπολογίας μπροστά σας, χωριστή, τροπολογία, χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος. Πρόκειται για την τροπολογία 79 της κυρίας Χάντζλικ. Υπέρ. Σηκώστε τα χέρια αν είστε υπέρ, παρακαλώ αν είστε υπέρ του πρώτου μέρους αυτής της τροπολογίας. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ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 Φτάνουμε στην νεοτολογική σκέψη τώρα. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 2. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τρία. Ε, με συγχωρείτε. 29. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Η τέσσερα απορρίπτεται. Η πέντε καταπίπτει. Η 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 32 προς 2 και 5 αποχές. Συγχαρητήρια Λουκά. Περνούμε τώρα στην επόμενη έκθεση, σημείο 16. Και πάλι γνωμοδότηση επί της ουσίας είναι υπεύθυνη η ΙΜΚΟ, ο ίδιος εισηγητής. Συμβάσει ψηνάτων που φορεί τα αστυνομία του τομεί του είδα του ενέργεια των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αρχίζουμε με τι τροπολογίε. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε το πρώτο, της πρώτη ψηφοφορία on block. 44, 45, 46 εγκρίνονται. Όχι. Ψηφίσαμε το πρώτο μπλοκ. 44, 45, 46. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Είστε κατά αυτή τη ψηφοφορία σαν μπλοκ. Εντάξει. Δεν ψηφίζουμε on block. Ας ψηφίσουμε Τι 44. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47. Όχι, θέλετε να κάνουμε παλήθευση ηλεκτρονικού 46. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση 47. Αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έχουμε λοιπόν ένα δεύτερο ψηφοφορία on block. Αν δεν είναι κανείς αντίθετος, ψηφίζουμε αυτό το δεύτερο block. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση του 54, αρχίζει η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64. Προφορική τροπολογία της κυρίας Ντεσαρνέζ. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι, την ψηφίζουμε. Και εδώ έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 65. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 67. Ε, αρχίζει ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 Συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 26. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τρι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Λίγη ψηφοφορία. 21 προς 5 και 4 ε, αποχές. Συγχαρητήρια. Ας πέρασουμε τώρα. Ας επιστρέψουμε τώρα στην αρχική σειρά, δηλαδή στο σημείο 11. Αυτή είναι μια διαδικασία συνένεση, είναι συμφωνία, είμαι εισηγητή. Συστήνω να δώσουμε τη συνένεση. Δεν υπάρχουν τροπολογίες, α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρόκειται για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Μολδαβία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Προτείνω λοιπόν στο πλαίσιο της διαδικασίας συνένεσης. Εγώ προτείνω στους συγητής να δώσετε την έγκρισή σας. Είναι διαδικασία έγκρισης. Κλείνει η ψηφοφορία. 29 υπέρ, 0 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Σημείο 12. Εδώ μιλάμε για ένα σχέδιο ε, εκθέση για τις διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας σταθεροποίηση και Σύνδεσης ΕΚ Σερβίας καθώς και της προσωρινής Συμφωνίας ΕΚ Σερβίας. Μιλάμε για νομοθετική έκθεση. Υπάρχουν οκτώ τροπολογίες. Ο εισηγητή είναι ο Γιούλιο Βίνκλερ από το ΕΛΚ. Α ψηφίσουμε ξεκινώντας από τις τροπολογίες. Τροπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 11 υπέρ κατά υπέρ, 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 12. Υ... Ας ελέγξουμε την τροπολογία 11, άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για την πρόταση της ε, Κομισιόν υπέρ Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 29 εναντί ε, μίας, καμία αποχή. Ε, για το ε, σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ξανά, άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέρμα ψηφοφορίας σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε το ίδιο λοιπόν αποτέλεσμα 29 υπέρ, μία ψηφοκατάκα, μια αποχή, συγχαρητήρια στον Γιούλιο Βίνκλερ. Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές μας, ο εισηγητής δεν θα μπει σε διαπραγματεύσεις για συμφωνία. Θα γίνει πλήρης ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Περνάμε στο αρχείο 13. Ερώτηση για προφορική απάντηση σε σχέση με τα μέτρα προστασίας της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγέ ναι, συνήθιστα χαμηλή τιμή από την Κίνα και ιδίως όσον αφορά τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες. Εισηγητής είμαι εγώ. Θα σας ενημερώσω ότι θα πρέπει να δώσουμε... Να αναφέρουμε τον Ντάνιελ Κάσπερη και τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις που συνεισέφεραν στη σύνταξη του ερωτήματος. Έχουμε ωστόσο 11 τροπολογίες. Ας ψηφίσουμε. Ας τις ψηφίσουμε. Συμβιβαστική 1 σε δύο τμήματα. Τρία τμήματα. Α, Ξεκινάμε την ψηφοφορία με μαζική ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Για την παράγραφο 5. Συγγνώμη, παράγραφο 4. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της παραγραφού 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 5 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και δεύτερο τμήμα παραγραφού 5 ε, Συγγνώμη, πρώτο τμήμα, ε, πέμπτη παραγράφου, 5, προηγούμενη ψηφοφορία ήταν ε, ψηφοφορία κατά τμήματα του πρώτου τμήματος παραγράφου 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τέλος, ε, περνάμε στο ε, τελευταίο κομμάτι της κατά τμήματα ψηφοφορίας, δεύτερο τμήμα, πρώτο τμήματος της παραγράφου 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρινέται με 28 ψήφους υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Περνάμε στο σημείο 14. Αυτή εδώ είναι μια διαδικασία έγκρισης το πρωτόκολλο στην Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ισραήλ για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ισραήλ σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων. Η γνωστή, το γνωστό πρωτόκολλο CAA. Εδώ έχουμε μια διαδικασία έγκρισης. Εγώ είμαι εισήγητη Το σχέδιο συστασίσμου, μου, όπως γνωρίζετε, είναι να μην δώσουμε συνένεση, να μην δώσουμε πλήρη συνένεση. Προτείνω δηλαδή να ανασταλεί η ψηφοφορία για δύο έτη. Α, ωστόσο υπάρχουν διάφορες τροπολογίες. Ξεκινάμε λοιπόν με τις τροπολογίες ωστόσο για να είμαστε σαφείς, οι πολιτικές ομάδες έχουν συμφωνήσει για τη διαδικασία ψηφοφορίας και για τη διασαφήνιση των πιθανών αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. Και έχουν συμφωνήσει σε ένα σημείωμα. Αναφέρομαι λοιπόν στο σημείωμα που υπάρχει στο αρχείο σας. Ας ψηφίσουμε λοιπόν για να δώσουμε τη συνένεση στο πρωτόκολλο. Ποιοι είναι υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας. Όσοι είναι κατά. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Πρέπει να ψηφίσουμε τώρα λοιπόν τις τροπολογίες. Τροπολογία 1 υπέρ. Ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ψηφίσουμε για το σχέδιο πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και κλείνει η ψηφοφορία. Και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως και με την πρώτη ψηφοφορία εγκρίνεται με 15 υπέρ, 13 κατά και δύο εποχές. Δεν δίνουμε συγχαρητήρια στον εισηγητή. η επεξηγηματική μου δήλωση θα αποσυρθεί επειδή έρχεται σε αντίθεση με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Περνάμε στο σημείο 17. Εδώ έχουμε μία γνωμοδότηση. Το σημείο 17 αφορά μία γνωμοδότηση για την ΑΦΕ, ε, μία ε, ΑΦΕΤ για τη Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Κεντρικής Αμερικής αφετέρου. Αυτή η συμφωνία σύνδεση, όπω γνωρίζετε, περιλαμβάνει μια πλήρη εμπορική συμφωνία. Εμεί, ωστόσο, εδώ παραμένουμε μόνο ως νομοθετική επιτροπή. Η συζητητή μα είναι ο Παύλο Άλμπα. Κατά πόσο θα δώσουμε δηλαδή εδώ τη συνένεσή μας σε αυτή τη συμφωνία από την ΑΦΕΤ. Υπάρχουν 46 τροπολογίες για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Ξεκινάμε από αυτές τις τροπολογίες. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία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 από τον εισηγητή και τον πρόεδρο κάποια αντίρρηση για την προφορική τροπολογία καμία ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία την έχετε στα αρχεία σας αν δεν κάνω λάθος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά ε, καταπίπτει. Η 7, ας ελέγξουμε την 7 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Επανερχόμαστε δηλαδή στην τροπολογία 7 και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται συγγνώμη 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ 27 ε, συγγνώμη 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 4 κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τώρα σχέδιο γνωμοδότησης ε, στο συνολό της ε, άρχεται ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον Παύλο Ζαλμπά. Περνάμε στο σημείο. Ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την ΑΦΕΤ μια στρατηγική ψηφιακή ελευθερία στην εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 57... 57 τροπολογίε. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχέ. Επαναλαμβάνουμε. Α, ναι, ηλεκτρονικός έλεγχος. 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την συμβιβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται. Διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 8. Υπέρ. Α. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές δεκτή ηλεκτρονικός έλεγχος. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 21. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 22 και 23 και 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά κατά αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος, συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία, έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Συμβιβαστική 7α. Καταπίπτει. Τροπολογία 50 και 51 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 50-51. Άρχεται η ψηφοφορία. Και έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 55 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Δεκτή. 56 υπέρ. τα αποχές δεκτή. Γίνεται κάποιος διάλογος εκτός μικροφώνου. λέει ο πρόεδρος, όταν υπάρχει διαχωρισμένη ψηφοφορία, οι φιλελεύθεροι πάντοτε είναι νικητές. Έχουν τα ενία. Λοιπόν, τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο κομμοδότησης ως, ε, όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Και υιοθετήθηκε με 25 υπέρ, 4 κατά. Συγχαρητήρια στον συντάκτη. Επί της είναι η ΑΦΕΤ, ο Μπέρτ, Μπέρτ Λάγκε, είναι ο συντάκτης μας και είναι οι συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΙΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ε, για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας Ευρωπαϊκή ε, Ένωσης Καζακστάν. Έχουμε 26 και αρχίζουμε με την συμβιβαστική 1. Υπέρ, κατά, βοχές δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ κατά από... Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σας, ε, κασαρά να βλέπω. Ε, τρία, τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5, 6 και όχι, 5 και 6 μαζί, 5 και 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έντεκα. Έντεκα. Ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. όχι, 10 υπέρ κατά αποχές. Α, 12 λέει ο πρόεδρος τώρα, μάλιστα, συγγνώμη. 12 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Όχι, το 13 ε, ε, απορρίφθηκε, το 14 εγκρίθηκε. Αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 14, λέει ο πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Η 14 απερίφθη. Τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 16 Ε, είναι ε, ε, διαχωρισμένη ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 ηλεκτρονικά τη 17 άρχεται η ψηφοφορία Έληξε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεκτή, δεκτή. Με 18, η, η τροπολογία 18, υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα, ε, πέρας της Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικά τη συμβιβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. Η 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και η τελική ψηφοφορία Άρχεται, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία για το τροποποιηθέν ε, σχέδιο νομοδότησης, έλικες η ψηφοφορία εγκρίθηκε. 24 υπέρ, 2 αποχές, 3, 2 ε, κατά, 3 αποχές. Συγχαίρω των Μπέρντ Λάγκε. Σημείο 20. Είναι μια γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία. Ο Σαϊέτ Καμάλ είναι ο εισηγητή, ο συντάξη γνωμοδότησης, ενδιάμεση έκθεση ενόψη θετική έκβαση τη διαδικασία έγκριση κλπ. Έχουμε 26. Όχι, έχουμε, συγγνώμη, έχουμε 10. Ε, τροπολογία 1, περίφθη, τροπολογία 2, πρώτο τμήμα, υπέρ κατά αποχές δεκτή, δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές δεκτό, ε, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το πρώτο τμήμα παρακαλώ τροπολογίας 4 δεκτή παρακαλώ, παρακαλώ, ακολουθήστε τον κανόνα μου. Εάν υπάρχει δια, ξεχωριστή ψήφος, ακολουθήστε τους φιλελεύθερους. Αυτοί ανεβάζουν και κατεβάζουν βασιλείς. Λοιπόν, το, τώρα ψηφίζουμε. Τροπολογία 4, δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχισε ψηφοφορία, έληξε ψηφοφορία. 21 υπέρ, 3 κατά, 2 εποχές. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, στον Σαγιάρ Καμάρ. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύ πειθαρχημένη ψηφοφορία αυτή που πάντοτε είναι ένα δύσκολο μέρος ε, του, της ατζέντας μας. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Θα ήθελα λοιπόν, παρακαλώ ακούστε με. Ε, υπάρχουν άτομα στην αίθουσα I want the people with their faces looking at me, not their backs. Ε, ήθελα να βλέπω τα πρόσωπα των ε, προσώπων που είναι μέσα στην αίθουσα και όχι την πλάτη τους, λέει ο πρόεδρος. Item 21. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο 21. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Όπως ξέρετε, αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα για τις συνεχιζόμενες για το συνεχιζόμενο προκαταρτικό αν το πω έτσι στάδιο των διαπραγματεύσεων είναι διμερής ε, η ομάδα εργασίας είναι διμερής με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η ομάδα αυτή εξέδωσε μία προσωρινή έκθεση που και η τελική έκθεση θα υποβληθεί στο τέλος του χρόνου. Γι' αυτό αποφασίσαμε να παρέμβουμε και να αφήσουμε να το, την Κομισιόν και το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει επ' αυτού, όπως ξέρετε. Ζητήθηκε να από τον συντάκτη να, να ετοιμάσει μία, ε, ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, και τον έχω, ε, την έχω διατυπώσει και είναι στο φάκελό σας. Η... Συζητήσαμε με τα συμβαλόμενα μέρη και με την Κομισιόν και όταν ολοκληρώθηκε η, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, ακούσαμε και την άποψη των Αμερικανών ομολόγων μας ε, όταν ήταν στις Βρυξέλλες σε μια επιπλέον συνεδρίαση της ομάδα εργασία. Ο Μάρτι Κάλλας που είναι το διοικητικό στέλεχο υπεύθυνο για αυτό το φάκελο με βοήθησε ιδιαίτερα αλλά και οι συνάδελφοί μου από την πλευρά των ΗΠΑ επίσης για να συντάξω το σχέδιο γνωμοδότησης και ε, προφανώς βεβαίως ε, μπορεί να βελτιωθεί με τις τροπολογίες σας, δεδομένου ότι εδώ κάνουμε το, την πρώτη συζήτηση. Το, το αφήνω στα χέρια σας, αυτή τη γνωμοδότηση τώρα είναι στα χέρια σας για βελτιώσεις, για σχόλια, για τροποποίησεις κλπ. Ε, επικέντρωσα την προσοχή μου στα βασικά, στα κέρια σημεία της διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο εταίρων ε, και τονίζω ορισμένα συγκεκριμένα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να σας την παρουσιάσω. Περιμένω ότι τα σχόλιά σας δεν είναι πολύ μεγάλη δυναμοδότηση. Ε, προτίμησα την την ποιότητα, επικεντρώθηκα δηλαδή στην, στα πολιτικά θέματα. Ποιότητα και όχι ποσότητα. Και θα ήθελα να αρχίσω να, και να ακούσω τις απόψεις της μόνιμης Επιτροπής Εποπτείας Πρόεδρε. Μ' Έτσι, εντάξει, Ε, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Ήδη στο προσχέδιο του σχεδίου σας ε, συζητήσαμε όλοι μαζί, συμπεριλάβατε τις απόψεις μας, τις παρατηρήσεις μας, έτσι ώστε ήδη ε, ενσωματώσατε ορισμένες ε, τροποποιήσεις που ζητήσαμε. Τώρα, γενικές σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι υπάρχει μία βασική παρατήρηση, μία ένα βασικό θέμα. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και με τις γειτονικέ χώρες έχουν ορισμένες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα ή μήπως θα έπρεπε εμείς ως Ένωση εφόσον συνομιλούμε με, τους, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, να συμπεριλάβουμε και αυτά τα στοιχεία. Διότι για τις ε, εμπορικές εταιρικές μας σχέσεις έχει μεγάλη σημασία η διαμόρφωση των συνόρων και πώς ανοίγουν ή κλείνουν τα σύνορα των Πολιτείων προς τις γειτονικές χώρες. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα αυτό. Θα πρέπει ίσως να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Εάν αλλάζει κάτι μετά από αυτήν την νέα διάσκεψη ΑΠΕΚ η οποία έγινε. Μήπως σημειώθηκαν αλλαγές. Θέλω να προσθέσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως όλοι ξέρουμε, ε, βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο και Γι' αυτό δεν ξέρω εάν την τελική μας έκθεση πρέπει να την αναβάλουμε και να την υποβάλουμε μετά τις αμερικανικές εκλογές. Δεν ξέρω ακριβώ ε, ποια ημερομηνία γίνονται οι εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την θαυμάσια συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί βεβαίως ε, αυτές τις μέρες, αυτή τη βδομάδα και γραπτός θα υποβάλω εγώ αυτές τις δύο παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πράγματι, ήταν μεγάλη χαρά που συνεργαστήκαμε με, την, με το ΕΛΚ και αυτή η συνεργασία θα αποφέρει καρπούς θετικούς. Ο κύριος Σόλτς. Α, ο Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα απλά να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε και κύριε Εισηγητή για αυτή την καλή κίνηση που πιστεύω μας παρέχει αυτό το έγγραφο. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ώστε να άρουμε τους φραγμούς και να αυξήσουμε το ΕΠ και στις δύο πλευρές. Είναι μια ε, ευκαιρία κέρδους για όλους, καθώς και ευκαιρία μόχλευσης της οικονομικής μας εξουσίας και το βλέπουμε αυτό στις κοινέ προσπάθειες της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ενώπιον της Κίνα για τις Πανίσγες Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και σύμφωνα μαζί σα πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαπραγματεύση το συντομότερο δυνατόν το, στις του 2013 όπω προτείνεται και να προσπαθήσουμε να σημειωθεί η πρόοδο πριν από το τέλο τη θητεία τη τρέχουσα Επιτροπή. Θα ήθελα να σα αναφέρω τι δικέ μου προτεραιότητε ε, εκ μέρου τη ομάδα των Φιλελευθέρων, το να αυξήσουμε τη συμβατότητα των κανονιστικών καθεστώτων, δηλαδή καλύτερη ε, τυποποίηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμπεριλήφθη στην ημερήσια διάταξη και στην προηγούμενη ολομέλεια. Τον εξυγχρονίσουμε του εμπορικού κανόνε ε, για να ρούμε του τους νέου φραγμού. Αυτό είναι σημαντικό με τι νέε τεχνολογίε που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται. Η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόψη δικαιοδοσία και για τι εξωτερικέ πολιτικέ. και σκέφτομαι επίση και το cloud computing και τις κυρώσεις προς το Ιράν καθώς και το πώς θα επηρεαστεί η προστασία των δεδομένων μας. Ε, πιστεύω ότι όλα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις συζήτησή μας με τις ΗΠΑ όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Στο σχέδιο γίνεται εστίαση στην προστασία και την επιβολή, αλλά πιστεύω ότι επίσης θα πρέπει να έχουμε σαφείς απόψεις και εικόνα για το ρόλο που θα παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε, λαμβάνουμε όλο και περισσότερες ενδείξεις Όπω έγινε στι συζητήσει και στι ψηφοφορίε για το ΑΚΤΑ, ότι το τρέχον σύστημα δεν είναι βιώσιμο στην ψηφιακή εποχή και δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα που θα εμποδίζει τον εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες. Συνεπώς πιστεύω η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία είναι σημαντικό, καθώ και η διαχείριση των διανοητικών δικαιωμάτων. Υπάρχει κατακαιρματισμό και αυτό ε, είναι επιβλαβές για τις ευκαιρίες ε, για τις επιχειρήσεις ε, καθώς και τη συνεργασία μας με την εταιρική, και την εταιρική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της βελτιωμένης πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις όπως συζητήθηκε και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διακόψω εδώ προς το παρόν, αλλά προς το στη συνεχή μας συνεργασία και με την ε, αντιπροσωπή των ΗΠΑ σε αυτό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, επόμενος ο κύριος Στέρντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι κάνατε πολύ καλή δουλειά. Θέσατε τα θεμέλια για το μέλλον. Η ερώτησή μου προς την Επιτροπή είναι ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση. Αναμένουμε ουσιαστικά να ολοκληρωθεί επί παραδείγματι η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με τον Καναδά Έχουμε ξεκινήσει πλήρε διαπραγματεύσει μεταξύ τη Επιτροπή και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να μα δώσετε ω Επιτροπή μια εικόνα τη τρέχουσα κατάσταση. Θα μα βοηθούσε ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι είναι από τι πιο συναρπαστικέ προοπτικέ που έχω δει σε αυτό το κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι ευκαιρίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτέ τι διαπραγματεύσει είναι τεράστιε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ο κύριος Ντάρτμουθ Νομίζω ότι ο κ. Σούλτς είναι πρώτος. Ο κ. είναι πρώτος στη λίστα. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω επίσης εσάς για την εργασία σας, την ομάδα παρακολούθησης. Πιστεύω ότι εδώ η ομάδα παρακολούθησης ε, παίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των συζητήσεων στην Επιτροπή και στη συμμετοχή και ε, καλό όλα τα μέλη της Επιτροπής να συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Γενικά πιστεύω, συμφωνούμε όλοι, ότι αυτή η έκθεση αφορά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη συζητήσει στην Επιτροπή, στο παρελθόν κάναμε πολλές προσπάθειες να δημιουργήσουμε ένα εφοροσύγχρονο υπερατλαντικό πλαίσιο συνεργασία και ποτέ δεν πέτυχε. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να ζητήσω από όλους μας και από την Κομισιόν αυτό που θέλω να σα ρωτήσω πώ έχουμε, πώς είμαστε τόσο αισιόδοξοι ότι αυτή τη φορά θα καταλήξουμε σε θετικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε πρέπει να πατάμε καλά με τα πόδια μας στη γη, να είμαστε ρεαλιστές, να μην ε, υπερεκτιμάμε τα πράγματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο των διμερών διαπραγματεύσεων. Η ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου έχει έναν τίτλο δύσκολο θέση εργασίας και ανάπτυξη, αλλά πιστεύω ότι επικεντρωνόμαστε λίγο υπερβολικά στον ορισμό της ανάπτυξης και του ρόλου που θα παίξει το εμπόριο στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό δεν δείχνει επαρκώς την... Ε, σχέση αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ και ποιο είναι το πλαίσιο στην αγορά, στην αγορά εργασία ε, και πιστεύω ότι το πλαίσιο που χαρακτηρίζει αυτό το σχέδιο θα πρέπει να αποτυπώνεται κάπω καλύτερα. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο που τώρα με το σχέδιο έκθεσή σα έχουμε ένα πολύ καλό έγγραφο μπροστά μα, αλλά πρέπει να το εμπλουτίσουμε ώστε ω ε, βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορούμε να αποτυπώσουμε το πλαίσιο στο οποίο εμεί προωθούμε και καθοδηγούμε αυτή τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο ακόμη παρατηρήσεις. Το πέμπτο σημείο που αναφέρατε, ότι θέλουμε να έχουμε ολοκλήρωση της εσωτερικής ε, διατλαντικής αγοράς το 2015. Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό για τις γενικές ε, οικονομικές δραστηριότητες με τις υπόλοιπες χώρες, διότι σήμερα το iPhone, για παράδειγμα, παράγεται κατά 15% της αξίας του στην Ευρώπη, αλλά το 45% ήταν στην Κίνα. Τι σημαίνει λοιπόν για αυτή την εσωτερική αλυσίδα κατά κάποιο τρόπο εάν δεν ε, συμπεριλάβουμε, δεν λάβουμε υπόψη τις νέες εξελίξεις του διεθνούς εμπορίου στην έκθεση, παραμένουμε σκεπτόμενοι βάσει χαρακτηριστικών του παρελθόντος, συνθήκων του παρελθόντος. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αρχίσουμε να κατανοούμε ότι αυτή η διατλαντική συνεργασία θα πρέπει να αποτελέσει κομμάτι ενός πολυμερού συστήματος εμπορίου. Και με αυτό με οδηγεί στα σημεία 15 και 16. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο αιτήματα. Ναι, συμφωνώ. Χρειαζόμαστε να σκεφτούμε με νέο τρόπο το σύστημα εμπορίας ε, γενικότερα με νέους κανονισμούς, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον από κοινού με τις ΗΠΑ ε, θέσουμε κανονισμούς που θα αποτελέσουν κριτήρια, που θα θέτουν τα κριτήρια. Δεν είναι επαρκές. Ναι, από την αρχή πρέπει να πούμε ναι, ότι πρέπει να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία μαζί με άλλους να καταλήξουμε σε αυτούς τους νέους κανονισμούς. Να συνεργαστούμε για την εκπόνηση αυτών των κανονισμών. Και τέλος, ε, ίσως δεν το κατάλαβα καλά, αλλά νομίζω ότι αυτό που είχαμε συζητήσει την τελευταία φορά στην ομάδα παρακολούθησης, τα πρότυπα, ο νέος κοινό κανονισμός ε, για ορισμένους τομείς αναπτυξιακούς, επιστημονικούς, τεχνολογικούς πρέπει να ενοποιηθούν, να ομογενοποιηθούν διότι διαφέρουν και πρέπει να εστιαστούμε κάπως και σε αυτό υπάρχει ανάγκη για την οικονομική ανάπτυξη και οι δύο εταίροι που περιγράφουμε εδώ να συνεργαστούν έτσι για ε, πιο ε, πρόσφορη συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ και τώρα η ΕΦΔ, ο κ. Ντάρτμουθ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εκδηλώσω το ενδιαφέρον μου, ε, το συμφέρον μάλλον. Εγώ έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο μου και έχω ζήσει για αρκετά χρόνια ως ενήλικας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένω πολιτής του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έγινα Αμερικανός πολίτης, παρότι είχα την επιλογή. Θα έλεγα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια μεγάλη και πολύπλοκη χώρα δεσμευμένη για να εξυπηρετεί τα δικά της εθνικά συμφέροντα με μοναδικό τρόπο. Το εγχείρημα λοιπόν αυτό θα επιτύχει αν ένα συγκεκριμένος τομέας αποτελέσει τον τομέα εστίαση των προσπαθειών των συναδέλφων και της Κομισιόν. Αν χρειαζόμουν λοιπόν να επιλέξω έναν τομέα, θα επέλεγα την παράγραφο 13 του κειμένου σας που μιλάει για την αναγκή αντιμετώπιση της πλήρου αμοιβαιότητα τη δημόσια συμβάση με ειδικότερη εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με όλο το σεβασμό που έχω προς του αξιότιμου συναδέλφου αυτού του Κοινοβουλίου, Έχουμε, όπως γνωρίζετε, μια συνθήκη εμπορική με τον Καναδά που προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε και φυσικά η κοινή ιδέα πολλών συναδέλφων είναι να αντιμετωπίσουμε πολλά, κατά την άποψή μου, άσχετα ζητήματα σχετικά με το Τέσαν και το ΣΥΟ e που δυσχεραίνουν την υλοποίηση μιας τέτοιας συνθήκης. Εμείς είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο μια συνθήκη με τον Καναδά που υπάρχει από το 1933 μέχρι που τις γυρίσαμε την πλάτη το 1975. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Παροτρύνω λοιπόν όλους να εστιαστούμε σε έναν τομέα και αυτός το τομέας κατά την άποψή μου θα έπρεπε να είναι οι δημοσίες συμβάσεις. Έχω άλλη μια παρατήρηση που πιστεύω είναι πολύ σημαντική. Σε αυτή την παραγραφό Β λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΕ μοιράζονται κοινέ αξίε και παρόμοια νομικά συστήματα. Και αυτό ήθελα να το τονίσουμε. Δεν αληθεύει ακριβώς η υπηρετική Ευρώπη. Το νομικό σύστημα της Υπηρετική Ευρώπης γενικότερα βασίζεται στον κώδικα του Ναπολέοντα. Ενώ το αμερικανικό σύστημα βασίζεται στο common law. Η μόνη χώρα που έχει όχι παρόμοιο, αλλά ουσιαστικά το ίδιο νομικό σύστημα με τις ΗΠΑ είναι φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει το ίδιο νομικό σύστημα. Το ίδιο ισχύει για τη Σκωτία, είπε. Αλλά αυτή είναι λεπτομέρεια, κύριε Πρόεδρε. Δεν πιστεύω ότι αξίζει να διακόψει ένας πρόεδρος την ομιλία μου γι' αυτό. Ουσιαστικά έχουμε το ίδιο νομικό σύστημα βασισμένο στις ίδιες νομικές αρχές. Ε, ποια είναι η γενική τώρα ε, η ιδέα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα με πρόθεση να άρει το common law από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσπάθησα να προκαλέσω τον ενδιαφέρον άλλων μερών για αυτό και δεν τα κατάφερα, αλλά θα εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή εν συντομία την ευκαιρία. Προτείνω λοιπόν αυτή η παράγραφος B να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Και ίσως υπό την προεδρία σας, ε, τη γνώση που έχετε του συνταγματικού δικαίου, ίσως ε, να τα καταφέρετε, να είστε ο καταλληλότερος άνθρωπος για να το πράξει αυτό. Άλλες παρατηρήσεις, κύριε Μάρτιν, ήθελα να πω ότι το σκοτσέζικο σύστημα είναι εξαιρετικά διαφορετικό από το Ηνωμένο Βασίλειο και άξιζε τον κόπο. Ευχαριστώ. Οι επόμενοι ομιλητέ. Ο Μπέρτ Λάγκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μία θέση, διότι το παράθυρο για τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσει με τις Ηνωμένε Πολιτείε θα προχωρήσει με συγκεκριμένα βήματα μετά τις εκλογές. Και γι' αυτό πρέπει τώρα να ε, δούμε τι θέση θα πάρουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα ξαναδούμε βεβαίως εξελίξεις μετά τις εκλογές, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το παράθυρο των δυνατοτήτων που ανοίγει τώρα, που είναι ανοιχτό και γι' αυτό πρέπει η έκθεση αυτή να είναι ισχυρή. Έχουμε και οι δύο πλευρές ε, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα ε, και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η βελτίωση. Ε, έχουμε και εμπειρίες αρνητικές οι οποίες δεν μας επέτρεπαν στο παρελθόν να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά πρέπει πάντοτε κανείς να αφήνει ένα περιθώριο αισιοδοξία, να, μην να μην είναι ποτέ απόλυτος. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα θεματάκια τα οποία αναφέρεται πρόεδρε, τα σημεία 6 και 7 παραδείγματο χάρη. Πρόκειται για τους δασμούς, τα τελωνία και τις μη, ε, τα μη δασμολογικά εμπόδια στις συναλλαγές. Ε, πολλές φορές συζητούμε τον συνδυασμό ε, αυτών ε, των ε, δασμών και βλέπουμε προστατευτικές τάσεις από την πέρα του Ατλαντικού πλευρά. Παραδείγματο χάρη αυτά τα προσκόμματα εξαγωγών της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας προς τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι πολύ έντονα διότι σκοντάφτουν ας πούμε στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες δεν είναι αποδεκτές και συμβατές από την άλλη πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν αν μπορέσουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση ε, στις αγορές θα έχουμε επιτύχει ένα μεγάλο βήμα πρόοδου. Ευχαριστώ. Σαϊάτ Καμάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να μακρυγορίσουμε και όλη τη μέρα. Κάποιοι από εμά είμαστε στην Ουάσιγκτον το Μάιο για την ε, Ατλαντική Ευρωμάδα, για το δίκτυο Ατλαντικής Πολιτικής και μιλήσαμε με κάποια άτομα από την Αμερικανική Δίκηση και, και με κάποιους βουλευτές του Κογκρέσου. Κάτι το οποίο συμφωνήθηκε είναι ότι όντως υπήρξε συνένεση όντως για κάποια συμφωνία, αλλά τι είδος συμφωνία θα είναι αυτή. Κάποιοι έλεγαν ότι θα πρέπει να, είναι να, περιέχει, να έχει κανονιστικό περιεχόμενο, αλλά θα πρέπει μεικτή πολιτική και εμπορική συμφωνία και ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Εάν θέλουμε τώρα να προχωρήσουμε, θα πρέπει να αρχίσουμε από αυτό εμείς. Τι είδους συμφωνία θέλουμε και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Νομίζω ότι αναφέρεται κάποια θέματα που θα πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι να δούμε ένθεν και ένθεν τι θέματα θεωρούμε ε, σημαντικά. Τα εμπορικά, τα θέματα υγείας, τεχνικά, κάποια άλλα και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε ε, επίσης και στα πλαίσια της ε, συμφωνίες είπα Ιαπωνία. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε στους διάφορους τομείς να έχουμε εναρμόνιση και να είμαστε σίγουροι. Δεν θα αλλάξουν τα πράγματα και μετά κάποιοι μας στο πρόγραμμα. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε και να συνειδητοποιήσουμε και νομίζω το είπαν κάποιοι συνάδελφοι στις ε, ιστορικές, παραδοσιακές διαφορές τις οποίες έχουμε με τον τρόπο με τον οποίο τα διανοητικά δικαιώματα πίν τα αντιμετωπίζουμε βλέπουμε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θέματα του copyright, των διατονικών δικαιωμάτων, των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ε, την χάνουν πολλών συζητήσεων και ενδιαφέροντος, διαφορετικά από ότι ε, αντιμετωπίζει διαφορετικά από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην κάνουμε τυποποίηση και ε, εναρμόνιση Απλώ για να την κάνουμε. Δεδομένου ότι πολλέ φορές οι προδιαγραφές που ισχύουν και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν επίσης ε, θέματα όπως στον τραπεζικό τομέα που είναι διαφορετικά και σημαντικά για τους μεν και τους δε. Και δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εναρμόνιση. Υπάρχουν επίσης μηχανισμοί και μέσα πάρα πολύ πολύπλοκα το οποίο χρησιμοποιούνται και είναι διαφορετικά για τους Αμερικανούς και για μας. Τα διάφορα μετοδοτικά προϊόντα, Φερρυπίν. Επίσης, πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι υποστηρίζουμε τις πολυμερείς συμφωνίες και θεωρούμε ότι είναι υποδέστερες αυτών οι διμερείς. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι και αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε αντιληπτό και μας απασχόλησε τη διάρκεια των ε, ε, γύρω των συζητήσεων Ντόχα, είναι αυτό το οποίο ελέγχθη τότε να ανοίξουμε περισσότερο την πρόσβαση της ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει και εμείς να δούμε κατά πόσον αυτό ισχύει. Δηλαδή, δεν θα πρέπει και η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να φανούν ότι κάνουν συμφωνίες οι οποίες δεν θα είναι πάντα επωφελείς για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το προσέξουμε. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν στα θέματα τα εμπορικά και προβλήματα και υπάρχουν και τα δυναμικά τα οποία θα πρέπει ε, Εμεί να προσέξουμε. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια τέτοιου είδου συμφωνία, θα πρέπει να δούμε, επαναλαμβάνω πρώτα απ' όλα, τι είδου συμφωνία θέλουμε συγκεκριμένα, για να μην μακρηγορούμε και κάνουμε, κάνουμε γενικότητα. ευχαριστώ. Η Επιτροπή τώρα, παρακαλώ. Ο Ιγνάσιο Ρεβερσιέ είναι εδώ, ο οποίος είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό στον ε, Γενική Διεύθυνση Γνάσιο Γαρσίου, Λόγος, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με μεγάλη ευχαρίστηση θα μιλήσω για αυτή την τόσο σημαντική και επίκαιρη έκθεση. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι χαιρετίζουμε την έκθεσή σας που την παρετοιμάσατε με την ομάδα παρακολούθησης από κοινού πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την συμφωνία αυτή που θα είναι λεπτομεριακή και μεγάλη επίβολη και φιλόδοξη. Αρχίσαμε συζητήσεις με τις ΙΠΑ στην αρχή του έτους αυτούς. Ξέρουμε ότι τα πράγματα δεν ήταν δεδομένα, διότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ ημών και ημών ε, όσον αφορά την προσέγγιση για κάποια θέματα και πιστεύω ότι στην προσωρινή έκθεση μπορώ να πω ότι καταλήξαμε σε κοινή κατανόηση για κάποια θέματα με τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, ότι η πιο εποφελής προσέγγιση οικονομικής και πολιτικής πλευράς θα είναι μία ε, φιλόδοξη συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα θέματα. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση που υποστηρίξτηκε και από εσά. Και αναφέρθηκαν κάποια θέματα όπως οι δημόσιες αγορές. Πρόκειται ε, ε, οι δημόσιες προμήθειες. Νομίζω ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα σημαντικά θέματα σε αυτή τη συμφωνία και θα πρέπει να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στην Αμερικάνικη αγορά, όπως ξέρουμε. Ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα για τη ΣΥΠΑ και για ξέρω πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε εκ... Εκτός μιας τέτοιου είδους συμφωνίας δεν νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες να προχωρήσουμε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό Πιστεύω ότι αυτός είναι ο κανονικός τρόπος τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Επίσης, βλέπουμε ότι αυτή την προσέγγιση θέλουν επίσης να την υποστηρίξουν και είπα. Επίσης, στην έκθεσή σας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα τα ρυθμιστικά, τα κανονιστικά. Κυρίως παραγράφους 7 έως 9. Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με οικονομικά ωφέλη, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα διάφορα βήματα που πρέπει να κάνουμε ώστε να γίνει υποφελής αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν ακόμη ρυθμιστικές και κανονιστικές διαφορές. Το θέμα αυτό δεν μπορεί να το ε, εξετάσει με ευκολία. Δεν πιστεύω ότι σε τέτοιου είδους θέματα θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε παρά μόνο εάν έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία που θα, και προτάσεις συγκεκριμένες που θα μας κάνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τις δύο πλευρές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα καινούριο, το οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν σε προηγούμενες συμφωνίες και αυτό θα είναι η μεγάλη πρόκληση στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι το μήνυμα της έκθεσής σας για αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συνεργαστούμε τους Αμερικανούς για να δούμε με ποιο τρόπο θα οργανώσουμε την καλύτερη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε περιμένουμε από τα εμπλεκόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέλη να μας κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις και μετά θα περάσουμε σε μια διαδικασία ευρύτερης διαβούλευσης ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τα βήματα που θα μας επιτρέψουν να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα. Δεν λέω βεβαίως ότι θα μπορέσουμε όλες τις διαφορές να τις απαλείψουμε ένθεν και ένθεν του ωκεανού. Απλώς Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία είναι η κατάλληλη συμφωνία για να ε, αμβλύνουμε κάποιες διαφορές. Το επόμενο βήμα που προβλέπει η Επιτροπή είναι πρώτα απ' όλα προσπαθούμε σιγά σιγά ε, και ως το τέλος του έτους να παρουσιάσουμε την τελική μας έκθεση που θα επικυρώσει τις προσανατολισμούς, τους γενικούς που έδωσε η προσωρινή εκθεσή, δεδομένου ότι και οι δύο ξέρουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις φιλόδοξες διαπραγματεύσεις και είπα το επιθυμούν. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι η τελική έκθεση, επαναλαμβάνω, θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, την ίδια με την προσωρινή. Επίσης, εργαζόμαστε και στο εσωτερικό των υπηρεσιών μας, διότι αν θέλουμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις αρχές του επόμενου έτους, χρειάζεται να κάνουμε μια μελέτη αξιολόγησης των ε, επιπτώσεων, θα λάβουμε υπόψη σχετικές οδηγίες. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταθέσουμε τις σχετικές προτάσεις στις αρχές του επόμενου έτους και καταρχήν λοιπόν ο στόχος μας να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις την επόμενη άνοιξη πιστεύω ότι είναι εφικτός. Τέθηκε και μια ερώτηση για τον Καναδά. Προφανώς, ολοκληρώνοντας τις διαπραγματεύσεις τον Καναδά εφέτος, θα είναι κάτι το θετικό, διότι θα δώσει ένα ισχυρό μήνυμα και προς τους φίλους μας τους Αμερικανούς και κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε στις διαπραγματεύσεις τον Καναδά είναι θέματα τα οποία ούτως ή άλλως θα πρέπει και με τη διαπραγμάτευση με τη ΣΥΠΑ να τα χειριστούμε. Άρα αυτό που θα κάνουμε στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης των Καναδά θα αποτελέσει μια προπαρασκευαστική εργασία κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι θα μπορέσουμε μετά να αρχίσουμε με τις ΙΠΑ. Τώρα για τα διανοητικά δικαιώματα να κάνω ένα σχόλιο που αναφέρθηκαν από πολλούς συναδέλφους σας. Πρέπει να πω το εξής. Και η και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάρα πολύ υψηλού κανόνε για την προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων. Και συνεργαζόμαστε ώστε να έχουμε και υψηλού επίπεδου προστασία αυτών των ίδιων δικαιωμάτων και σε τρίτε χώρε. Υπάρχουν διαφορέ βεβαίω στην ε, νομοθεσία και Βεβαίω, δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι μια τέτοιου είδου γενική συμφωνία θα αποτελέσει τον κανόνα ή τη βάση, ή το θεμέλιο επίλυση όλων των διαφορών σε αυτό το τομέα ή την εναρμόνιση. Πώς θα χειριστούμε αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο το συζητούμε με τους συναδέλφους για να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη προσέγγιση στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης. Και τελικά Απλώς και μόνο να πω ότι χαιρετίζουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαπραγμάτευση, διότι θα είναι πολύ σημαντικές και με γεμάτες προκλήσεις και η ομάδα παρακολούθησης και εποπτείας πάντα θα σας ενημερώνει για το τι ακριβώς γίνεται, κυρίως όταν αρχίσει όλη η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Μας ενδιαφέρει επίσης να δούμε Ποιες είναι οι δραστηριότητες που σκέφτεστε εσείς να αναπτύξετε με το Αμερικανικό Κογκρέσο και τους ε, εκεί συναδέλφους σας και η σχέση την οποία αναπτύσσετε εσείς είναι σημαντική για μας. Τελικά ένα σχόλιο για το μεγάλο θέμα γιατί τώρα μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι από ό,τι στο παρελθόν Πιστεύω ότι υπάρχουν τρία στοιχεία αυτή τη στιγμή τα οποία δεν είχαμε στη διάθεσή μας στο παρελθόν. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αναντήρητα μεγάλη πολιτιστική υποστήριξη, πράγμα που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δώσει ένα πάρα πολύ σαφές μήνυμα, πράγμα το οποίο σε πολιτικό επίπεδο δεν συνέβαινε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν. Επίσης, κατανοούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θα υποστηρίξει αυτή την πάρα πολύ σημαντική συμφωνία, αλλά και από την πλευρά των ΗΠΑ πρέπει να πω ότι είχαμε πάρα πολύ σαφείς ενδείξεις ότι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο έχει μεγάλη πολιτική υποστήριξη. Δεν πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει ε, έλλειψη υποστήριξη και από τη ΣΥΠΑ και καταλαβαίνουν ε, από οικονομική πλευρά ότι και είπα ότι όσο και σημαντική από οικονομικής άποψης να είναι μια οικονομική συμφωνία, εάν είναι διατλαντική είναι ακόμη πιο σημαντική. Και πιστεύω ότι με την ύπαρξη κοινών κανόνων σε διεθνές επίπεδο μπορούμε να προχωρήσουμε. Τελικά, Υπήρχε αντίληψη στο παρελθόν ότι οι διμερείς ε, διαπραγματεύσει ταξί ΕΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαν ε, αρνητικές επιπτώσει στο επίπεδο των συζητήσεων στο χείρο της Δόχα. Δεν ε, υπάρχει πλέον τέτοιου είδου θέμα. Ξέρουμε ότι ούτω ή άλλω υπάρχουν δυσκολίες σε επίπεδο γύρου διαπραγματεύσεων των, της Δόχα. Αντιθέτω το να λανσάρουμε μια τέτοιου είδου ε, φιλόδοξη διαπραγμάτευση μεταξύ ΕΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει σινιάλο και προ τρίτε χώρε ότι είμαστε ε, σε πολύ κοντά στο επίπεδο το να κάνουμε πολυμερεί διαπραγματεύσει, αλλά προσδίδουν και μεγάλη σημασία αυτή την τόσο σημαντική διμερή διαπραγμάτευση. Γι' αυτό έχουμε λόγο να είμαστε, όπω σα είπα, αισιόδοξοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν θα είναι εύκολα, το γνωρίζουμε όλοι θα πρέπει να χειριστούμε κάποια πάρα πολύ πολύπλοκα θέματα, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένω να ολοκληρώσουμε την πράγματα το 2014. Ναι, ενδεχομένω, αλλά πάντα δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η ουσία και το περιεχόμενο είναι πιο σημαντικέ από τις προθεσμίες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και χαιρετίζουμε και πάλι την έκθεσή σας. Ευχαριστώ.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 Είναι, είπε ο Πρόεδρος, συγγνώμη. Ε, ε, η πιο σημαντική συμφωνία αυτή, ε, την οποία έχουμε εμπλακεί για την ανάπτυξη και την εργασία, την απασχόληση και ευχαρίστησε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τα θετικά του σχόλια. Λοιπόν, με ορισμένες λίγες εξαιρέσεις, η υποστήριξη μιας φιλόδοξης διαπραγμάτευσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ ΕΕ υπάρχει. Υπάρχει στήριξη, υπάρχουν βάσιμες ε, ενδείξεις για με ένα πολύ καλό δυναμικό βελτίωσης και πρέπει να δείξουμε μια ισχυρή θέση. Ε, η προϋπόθεση είναι ε, να είμαστε, όχι θα έλεγα απόλυτα σίγουροι, αλλά αρκετά σίγουροι ότι δεν θα αποτύχουμε. Δεν πρέπει να πάμε με, μια, με ένα πνεύμα ητοπάθειας ε, στη διαπραγμάτευση, διότι οι συνθήκες είναι σκληρές, η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή και για να επιτύχουμε στο τέλος, για να ε, ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να καταπιούμε μερικά πικρά χάπια. όχι μόνο η αμερικανική πλευρά, αλλά και εμείς. Παραδείγματο χάρη στι δημόσιε συμβάσει, στι δημόσιε προμήθειε, στον αγροτικό τομέα, στις γεωγραφικές ενδείξεις, στις προδιαγραφές ε, των οχημάτων, της αυτοκινητοβιομηχανία. Αναφέρω ορισμένα καυτά ζητήματα όπου ίσως και εμείς να πρέπει να καταπιούμε το πικρό χάπι εξαρτάται ακριβώς από την ισορροπία την, την οποία μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τώρα, τι άλλες συμφωνίες πρέπει να εξετάσουμε. Όταν ζούσε ακόμα η Ντόχα, Ε, εξετάζαμε και άλλες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φιλόδοξες, αλλά σκοντάφταμε μονίμως τα προσκόμματα σε εμπόδια, σε εμπορικά εμπόδια, διότι δεν είναι μόνο οι δασμοί εμπόδια, υπάρχουν και άλλα εμπόδια, άλλης φύσεως δηλαδή, μη δασμολογικά. Άρα λοιπόν δεν μας αφορά μόνο η πρόσβαση στην αγορά, αλλά και οι κανόνες. Όπως ξέρετε, οι κανόνες πρέπει να συνάδουν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και πολλές φορές ο ΠΟΕ δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του, διότι επιδιώκει να εκδώσει ε, διεθνείς κανόνες, αλλά σκοντάφτει στα προσκόμματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει και οι Ηνωμένε Πολιτείε να εφαρμόζουν γενικά αποδεκτούς κανόνες, λογικούς κανόνες ε, και εμείς να δείξουμε μια καλή διάθεση. Αλλά πάντοτε να γνωρίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που παρουσιάζονται, οι οποίες πάντοτε υπερβαίνουν απλώς το πρόβλημα της, της πρόσβασης στην αγορά. Όποτε διαπραγματευόμαστε με τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι προκλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από μόνο την πρόσβαση στην αγορά. Ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ας πούμε ευαισθησίες εναντίον μιας συμφωνίας. Πολιτικά εμπόδια δεν υπάρχουν. Έχουμε την συμφωνία, την εταιρική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία έχει εγκριθεί από πολιτικής απόψεως. Οπότε αυτές είναι οι γενικές γραμμές με τις οποίες θα προχωρήσουμε και θα προσεγγίσουμε αυτή την γνωμοδότηση, αυτή την έκθεση. Είναι η πρώτη φορά που μια τόσο σοβαρή έκθεση θα εκδοθεί που θα καλύπτει την διαπραγματευτική μας γραμμή, το διαπραγματευτικό μας πλαίσιο με το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό εμπορικό εταίρο Γι' αυτό πρέπει να δηλώσω σαφώς την Κομισιόν ότι ό,τι λέμε το εννοούμε. Πριν ληφθεί απόφαση θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ και ε, με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα την Κομισιόν να δηλώνει ότι χαιρετίζουν την πρωτοβουλία μας και θα λάβουν υπόψη τις θέσεις μας. Περιμένω τις ε, τροπολογίες σας και θα επανέλθουμε βεβαίως στη συζήτηση των τροπολογιών και εν συνεχεία στη ψηφοφορία. 21 Σεπτεμβρίου το, στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Τελευταίο θέμα σήμερα το πρωί είναι η το ενωσιακό θελωνιακός κώδικα. Ε, ε, επί τη ουσία η επιτροπή είναι η ΙΜΚΟ. Ε, η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι ε, η κυρία Μουσκαρδίνη από το ΕΛΚ. Τα τελωνία θα πρέπει να είναι δική μας αρμοδιότητα και όχι τη ΣΥΜΚΟ, αλλά έτσι αποφασίστηκε στο παρελθόν, οπότε πρέπει να κινηθούμε μέσα στις αρμοδιότητές μας και να εκδώσουμε γνωμοδότηση. Και δίνω το λόγο στην ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία για να υποστηρίξω το ότι θα ήταν απαραίτητο να συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτό το ζήτημα αρμοδιοτήτων μεταξύ εμάς και της ΣΥΜΚΟ διότι αλλιώς θα συνεχίσει και στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Δεδομένων αυτών και ότι έχει περάσει η ώρα, έχουμε μιλήσει για το ζήτημα αυτό σε διάφορες ευκαιρίες. Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία αγορά και ενωμένη αγορά χωρίς εναρμονισμένο τελωνιακό σύστημα. Αυτή τη στιγμή ο τελωνιακός κώδικας που είχε ήδη αναθεωρηθεί πριν από λίγο καιρό χρειάζεται νέες μικρορυθμίσεις και ε, εξυγχρονισμό. Δυστυχώς, το σχεδίο που παρουσίασε η Κομισιόν δεν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή δεν μας ικανοποιεί εμάς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή διότι δεν συνάδει με τα όσα έχουμε υποστηρίξει σε διάφορες ευκαιρίες δηλαδή το πρόβλημα της πραγματικής εναρμόνισης το πρόβλημα των χρόνων εδώ έχουμε το 2020, έχουμε μπροστά μας 7 χρόνια χάος και δεν αντιμετωπίζει ούτε καν α, τους διαφορούς όρους που πρέπει να είναι ίδιοι σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Τους όρους κατανομής των δασμών. Εμείς ως Κοινοβούλιο Αυτέ τις υποθέσεις για το μέλλον εναρμονισμού των τελωνίων στην Ευρώπη, τα υποστηρίζουμε. Αλλά ενώ παραμένουν διάφορα προβλήματα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα δικά μας τελωνία, δηλαδή τα εσωτερικά μας τελωνία, τα τελωνία αγαθών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν στα δικά μα σύνορα τον ίδιο τύπο ελέγχων. Οι έλεγχοι δεν είναι οι ίδιοι, δεν δίδεται η ίδια προσοχή στην παραποίηση δεν προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο τόσο η εισαγωγή όσο και η αποστολή εμπορευμάτων. Εάν σε αυτό προσθέσουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με τις τροποποιήσεις και τη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Κώδικα που παραπέμπει στο 2020 η Κομισιόν, έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά βήματα ως Κοινοβούλιο για να παροτρύνουμε την Κομισιόν να έχει μια στάση πιο υπεύθυνη στη σημερινή Ευρώπη των 28 που αντιμετωπίζει μια κρίση η οποία εξαρτάται επίσης και από ένα εμπόριο και από αγορές που δεν προσαρμόζονται πλέον στις απαιτήσει μας. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε προηγουμένως τα προβλήματα του διεθνούς εμπορίου, ότι δεν συνάδει πλέον με τις απαιτήσει. Στην περασμένη του θητεία το Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει τροποποιήσεις και βελτιώσεις, αλλά κανείς ακόμη δεν έχει λάβει υπόψη. Δεν μιλάω μόνο για τα θεσμικά πρόσωπα στο πλαίσιο του εμπορίου, αλλά μιλάω και για, τους ευρωπαϊκούς, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οι λύσεις για τα κρίσιμα προβλήματα είναι λανθάνουσες. Και μέχρι να ξυπνήσουν ε, έχει περάσει πια ο χρόνος. Γι' αυτό το λόγο εμείς παρουσιάσαμε ένα κείμενο για το οποίο συμφωνήσαμε με τους συναδέλφους. Έχουμε τροπολογίες που υποβάλαμε σε σχέση με αυτό το κείμενο εγώ ίδια Δεσμεύομαι να παρουσιάσω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις μες στις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό το λόγο ζητώ από τους συναδέλφους να εκτιμήσουν και να υποβάλουν οτιδήποτε θεωρούν σημαντικό και ωφέλιμο ώστε να τροποποιήσουμε προς το καλύτερο την πρόταση της Κομισιόν η οποία αφενός κινείται προς την κατεύθυνση του, του επίγοντος και της ανάγκης χρειάζεται μια πρόταση. Δηλαδή, από την άλλη μας απογοητεύει, διότι ο επίγον χαρακτήρας μεταφράζεται σε αργοπορία και οι αποφάσεις δεν είναι τόσο οριστικές και κατάλληλες όσο θα θέλαμε. Ευχαριστούμε Κριστιάνα, Σκιώδης, κύριε Σούστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα ήθελα να πω ότι υπάρχει κίνδυνος να πρέπει να διορθώσουμε είτε μέσω τροπολογιών στην Επιτροπή ΙΝΤΑ είτε γενικότερα στην ΙΜΚΟ λαμβάνεται υπόψη ότι καλό θα ήταν να αναλάβουμε εκ νέου εμείς τις δικές μας αρμοδιότητες. Υπάρχει κίνδυνος αυτή να αποτελέσει μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Η αναδιατύπωση του τελωνιακού κώδικα σε εποχές κρίσης όπως σήμερα, σε εποχές όπου πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στον κόσμο, θα έπρεπε να φέρει την ίδια την Ευρώπη και του ευρωπαϊκά όργανα να μεταρρυθμίσει ε, ολοκληρωτικά με κανόνες που θα ευνοήσουν τις ε, συναλλαγές, την προστασία των διενωτικών δικαιωμάτων και που θα ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα και στον κόσμο και στην Ευρώπη. Κάποια στοιχεία μας ανησυχούν. Το πρώτο είναι οι υπερβολικές αναθέσεις εξουσιών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσω αυτού του μέσου τι στερείται το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις εξουσίες του σε σχέση με την Κομισιόν, με τις κατευθυντικές πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε μέχρι βάθους ποιο είναι το όριο ώστε να αποφύγουμε να υπάρχει υπερβολική εκχώρηση εξουσιών για σημαντικά ζητήματα, όπω για παράδειγμα οι κανόνε προέλευση. Το δεύτερο ερώτημα είναι η εναρμόνιση εσωτερικά. Ο τελωνιακό κώδικα σίγουρα αφορά τι σχέσει με το εξωτερικό, αλλά εμεί γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένο τρόπο αξιοποίηση των μέσων που μα προσφέρει η νομοθεσία για να ελέγχουμε τα λιμάνια τις προσβάσεις, ε, να εφαρμόζουμε τους δασμούς, να ορίζουμε τις κυρώσεις, είναι μια θεματική που απαιτεί εναρμόνιση πλήρη. Χωρίς αυτήν υπάρχει κίνδυνος ε, να επιτυχάνουμε αποτελέσματα επί χάρτο, αλλά ουσιαστικά πρακτικά να μην καταφέρουμε να επιτυχάνουμε αυτό το σύστημα ελέγχου που θα προστατεύει τους καταναλωτές μας και το δεγονιστικό μας σύστημα. Το τρίτο σημείο που δεν αντιμετωπίζεται και που θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με τροπολογίες ad hoc είναι ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση για να οριστεί καλύτερα το ζήτημα της ανεχνευσιμότητας, της ειχνηλασιμότητας. Αφενός δηλαδή θέλουμε να προστατέψουμε τους καταναλωτές 100% ε, και ε, αφετέρου δεν υπάρχει συνοχή στον τελωνιακό κώδικα. Δεν υπάρχει κάτι που να μας λέει πώς θα μπορούμε να ε, οριοθετήσουμε την ειχνηλασιμότητα. Εάν σε αυτό προσθέσουμε την παράλογη ε, σιωπή, για τις σημάνσεις των προϊόντων που εισάγονται στην Ευρώπη, όπως έχει ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια, έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο σίγουρα δεν είναι αισιόδοξο. Έτσι λοιπόν είναι δικός μας ρόλος ως κοινοβουλευτικού θεσμού να εργαστούμε για να βελτιώσουμε αυτό το κείμενο και ελπίζω ότι οι εργασίες και τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου θα βρουν ανταπόκριση και στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σιλβάνα Κοχμέριν, παρακαλώ. Thank you very much. Um, äh, σε αυτό το θέμα ε, υπάρχει μια κλασική αντιμετώπιση όπου όλοι εντός και εκτός Ευρώπης πιστεύουν ότι βεβαίως εδώ η Ευρώπη πρέπει να συμπεριφερθεί ομοιόμορφα, να έχουμε κοινά στάνταρτς, κοινή προσέγγιση, εναρμονισμένες διαδικασίες και αυτή ήταν και η αρχική πρόθεση. Έχω τώρα μία επιφύλαξη μετά από την ε, υιοθέτηση της ατζέντα της ε, Λισαβόνας και αφού λίγο την παραμερίσαμε, δεδομένου ότι έθετε μια χρονική προθεσμία, ε, δεν πέτυχε τόσο πολύ στους στόχους της στην τον ε, εκμοντερνισμό, ας πούμε, στην, ε, τον εξυγχρονισμό των ε, τελωνίων, του τελωνιακού καθεστώτος κλπ. καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ήταν ένα φιλόδοξο, σωστό σχέδιο που είχαμε, αλλά απέτυχε διότι υπάρχουν αυτές οι πολύ μεγάλες ή τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και στις αρμοδιότητες αλλά και στην βούληση ε, να επιφέρουν αυτόν τον εξυγχρονισμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο ε, πιστεύω ότι πρέπει να εμείνουμε, να προσεγγίζουμε φιλόδοξα ε, το σχέδιο αυτό, το χρονοδιάγραμμα βεβαίως να είναι ρεαλιστικό και να το δεχθεί ως ρεαλιστικό η Κομισιόν, αλλά να παραμείνουμε φιλόδοξοι, να επιμείνουμε και να επικρίνουμε σαφέστατα εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έδειξαν καμία διάθεση να προχωρήσουν με τον εξυγχρονισμό και τελικά κολυσιεργούν την πρόοδο. Κατά τα άλλα, εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξεις δεδομένου ότι εδώ αυτό συνάδει με το δικό μας ρόλο και ε, έτσι θα μπορέσουμε και να ελέγξουμε το τι γίνεται. Αυτά τα οποία προβλέπει η Κομισιόν, δηλαδή το εύρος της κάλυψης των κατεξουσιοδότηση πράξεων για μένα είναι προβολικό, διότι μετά ως Κοινοβούλιο εμείς έχουμε λίγες δυνατότητες να παρέμβουμε και να ελέγξουμε πλήρως. Γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε να είναι το εύρος αυτό ε, λογικό, να μην είναι υπερβολικά μεγάλο για να μπορούμε και εμείς να παρακολουθούμε. Άλλοι συνάδελφοι είπαν και ευχαριστώ ιδιαίτερα την ε, συντάκτρια ε, για την γνωμοδότησή της και για τις επικρίσεις και τα σχόλια τα οποία περιέχει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στέρντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώ εκ μέρους της ε, κυρίας Μακλάρκιν, η οποία είναι σκιώδης εισηγήτρια και δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ, αλλά μου, ε, μου ζήτησε να μιλήσω εκ μέρους της, δεδομένου ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική γνωμοδότηση εκ μέρους της ε, ΙΜΚΟ. Η κυρία Μακλάρκιν ε, ευχαριστεί την συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Μουσκαντίνη. Και πιστεύει ότι η Επιτροπή μας ακολουθεί ε, τη βασική προσέγγιση της επί Επιτροπής και ότι αυτή η γνωμοδότηση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον τελωνιακό κώδικα. Όπως λέει η συγγήτρια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ε, διαφερομένων και η διασφάλιση του νόμιμου ε, εμπορίου και η καταπολέμηση των παραχαραγμένων προϊόντων και των ε, προϊόντων μαϊμούδων η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών συμφωνεί με ε, αυτές τις βασικές γραμμές. Θα πρέπει να όμως να δοθούν ε, συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ρήτρες εξαιρέσεων σε ορισμένα κράτη-μέλη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη στην αποθήκευση δεδομένων με, με, μέσα τα οποία δεν είναι ηλεκτρονικά. Πρέπει να δοθούν ορισμένε ρήτρε εξαιρέσεων. Δεδομένου ότι ε, ορισμένα κράτη-μέλη λόγω τη ε, χρηματοοικονομική κρίση ε, έχουν προβλήματα στην ενσωμάτωση τη επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρονικά, στην πλήρη μηχανογράφηση δηλαδή. Και επίση θα πρέπει να ε, διευκολύνουμε τον ε, τελωνιακό κώδικα με την υιοθέτηση κοινών κανόνων που θα επιτρέπουν την αμεβαία αναγνώριση των κανόνων ε, και τη συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας των ενδιαφερομένων του κλάδου. Κατά τα άλλα υποστηρίζει την γνωμοδότηση και ευχαριστεί τη συντάκτρια. Ο πρόεδρος, ο, ο, ο, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τους προλαλήσαντες συναδέλφους ότι αυτή είναι μία ε, πρόταση την οποία επεξεργάστηκε πολύ σωστά η κυρία Μουσκαρδίνη. Θέλουμε όλοι να συμπλέψουμε, πρέπει όμως να προσέξουμε ποια είναι η, η, η, αρχική θέση της ΙΜΚΟ εμείς συζητούμε τώρα τον εξυγχρονισμό του τελωνιακού συστήματος κάτω από συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης και θα πρέπει να, να λάβουμε υπόψη και τις απόψεις των κρατών της Ευρωζώνης αλλά και εκτός της Ευρωζώνης γιατί εμείς θέλουμε βεβαίως να ισχυροποιήσουμε τη θέση της Ευρωζώνης αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και ε, την κατάσταση των σχέσεων με εκτός, ε, τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Γι' αυτό θα έλεγα, η, η με τις, τους σκιώδεις εισηγητής να ξανακαθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν ποια είναι τα βασικά στοιχεία από τα οποία ξεκίνησαν, πού βασίζονται ακριβώς οι βασικές τους απόψεις και πού είναι οι τα δύσκολα κομβικά σημεία λόγω της περιπλοκότητας του θέματος. Γι' αυτό ε, θέλουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ποιοτικά το περιεχόμενο της γνωμοδότησης και είμαι πρόσφυγος να συμμετάσχω σε αυτές τις συζητήσεις. Γενικά ευχαριστώ τη συντάκτη γνωμοδότηση για την εργασία της. Ο Πρόεδρος. Η Επιτροπή έχει τίποτα να προσθέσει. Ο κ. Τζιλίνσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζηλίνσκι. Διευθυντής τη Ταξούντ για θέματα τελωνιακής πολιτικής. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι εκτιμούμε πάρα πολύ την έκθεση και την δουλειά που έχει επιτελεστεί και τις απόψεις και το όραμα που εκφράζεται, που ευθυγραμμίζεται με τις απόψεις τι δικές μας στην ε, Ταξούντ και στην Επιτροπή γενικότερα θα έλεγα. Υπάρχουν πολύ καλές ιδέες, κάποιες από τις οποίες είναι πράγματι επαναστατικές και με μεγάλη ευχαρίστηση θα τις επεξεργαστούμε. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η εναρμόνιση ήταν ο στόχος μας. Η εναρμόνιση και η ενιαία εφαρμογή του ελληνιακού Κώδικα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε πόσο το θέμα των ε, τελωνίων είναι σημαντικό και άλλους τομείς. Προστασία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Ε, αποτροπή εισαγωγής επικίνδυνων και άλλων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΚΑΠ επίσης έχει σχέση. Η εναρμόνιση, εναρμόνιση λοιπόν είναι ο στόχος μας και θα πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Και βεβαίως θα πρέπει να προσθέσω ότι βεβαίως έχουμε περιορισμένες εμβέλειας ε, φιλοδοξίες ή δυνατότητες να ενεργήσουμε μάλλον, δεδομένου ότι είμαστε στα πλαίσια της ε, αναδιατύπωσης αυτού του νέου τελωνιακού πράγμα το οποίο είναι κοινή δουλειά μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Και η αναδιατύπωση είναι θέμα διαθεσμικής συμφωνίας που υπόκειται σε κανόνες που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε. Διαφορετικά θα αποτύχουμε να Έχουμε έτοιμο το νέο αυτό κώδικα πριν από τις 24 Ιουνίου 2013. Και δεν θα μπορέσουμε να τον εφαρμόσουμε με το σωστό τρόπο. Και αν δεν μπορέσουμε θα έχουμε τον παλιό, χωρίς ε, τη δέουσα νομική βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η αναδιατύπωση έγινε αποδεκτή και συζητήθηκε πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά στην ΙΜΚΟ έχει τρεις στόχους. Αναβολή εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης, διότι τα συστήματα πληροφορικής είναι πάρα πολύ δαπανηρά και δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να τεχθούν σε εφαρμογή πολλές φορές έγκαιρα. Δεύτερον, ευθυγράμμιση με την συνθήκη της Λισαβόνας. Τρίτος, για την αναδιατύπωση, ρυθμίσεις, διορθώσεις, γιατί πάντα υπάρχουν κάποια σφάλματα και θα πρέπει να βάλουμε υπόψη και το ε, νομικό σύστημα και πλαίσιο το οποίο αλλάζει πολλές φορές. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, μας περιορίζει ακόμη και ίδιος ο ορισμός της αναδιατύπωσης. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ειδικά θέματα. Ίσως όχι πιο σημαντικά. Εδώ όμως τέθηκε το θέμα των προσωρινών ε, παρεκκλήσεων και εξαιρέσεων σε θέματα IT. Υπάρχει το θέμα της δυνατότητας παράδοσης στα πλαίσια της IT. Αλλά υπάρχουν και χώρες που δεν προβλέπουν μια τέτοια διαδικασία. Φερρυπίν. Οι χώρε που δεν έχουν πρόσβαση, που δεν έχουν θαλάσσια σύνορα, πρόσβαση στη θάλασσα, δεν χρειάζεται να κάνουν και να αναπτύξουν ειδικέ διαδικασίε όσον αφορά τα ε, θαλάσσια σύνορα και την ε, σημασία των τελωνίων. Και πολλές φορές σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οι πράξεις που γίνονται είναι πολύ λίγες ετησίως. Άρα ε, θεωρείται η αλλαγή του IT πολύ δαπανηρή. Τώρα, διαβάζω τις σημειώσεις μου. Ο εξυγχρονισμός και η εναρμόνιση. Πιστεύω ότι η πρότασή μας είναι πάρα πολύ καλύτερη από τον παρόντα τελωνιακό κώδικα. Θέλουμε να προχωρήσουμε εμείς στην Επιτροπή πολύ περισσότερο. Ένα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησε για τα stumbling blocks. Έτσι τουλάχιστον μεταφράστηκε. Που μας μπλοκάρουν. Αλλά η κατάσταση στον τομέα αυτό είναι διαφορετική για τον καθένα. Πρέπει να βρούμε όμως τον κοινό παρανόμαστη ο κοινό παρανομαστή. Αυτά που μας ενώνουν είναι αυτά για τα οποία μπορούμε να συνενέσουμε και θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η ανάθεση και οι πράξεις εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μιλούμε για ανάθεση εξουσιών αρμοδιοτήτων, αλλά για ευθύνη. Μπορεί κάποιος να έχει την εξουσία, τη δύναμη να αναθέσει κάτι σε κάποιον, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι η ευθύνη. Λοιπόν, η ανάθεση ε? και η εφαρμογή είναι σημαντική. Και εδώ μπαίνει το θέμα της ευελιξίας. Βα... Καταλαβαίνουμε ότι το βασικό θέμα είναι θέμα το οποίο είναι ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ανάθεση και η ευθύνη που δίδεται για την εφαρμογή είναι επίσης σημαντικό. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι η ευθύνη. Ο κόσμος αλλάζει, έχουμε... It's easier Οι πράξεις εξουσιοδότησης επίσης είναι σημαντικές η βασική πράξη, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις διεθνείς συμβάσεις και τις ε, συμφωνίες ελεύθερου Μπορείου και γενικότερα το νομοθετικό πλαίσιο. Και ξέρουμε ότι κάποιες λεπτομέρειες που υπάρχουν στην βασική πράξη δεν μπορούν να μεταφερθούν στην, ε, στο επίπεδο των ε, διεθνών συμφωνιών, διότι χρειάζεται χρόνος για να περάσουν οι διαδικασίες από τα τρία θεσμικά όργανα, να γίνει ο τριμερής διάλογος κτλ. Δεν χρειάζεται να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, απλώς επαναλαμβάνω ότι η... όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα ευθύνης και ευελιξίας. Ολοκληρώνοντας, θα πω ότι εκτιμούμε τις ιδέες που συμπεριλαμβάνει την εκθεσή σας, θα πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε, αλλά όπως ξέρετε μας δεσμεύει το νομικό πλαίσιο και οι χρονικοί περιορισμοί, δεδομένου ότι είμαστε στην αναδιατύπωση σε αυτή τη φάση. Κυρία Μουσκαρντίνη. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω φυσικά όλους τους συναδέλφους για τη διαθέσιμότητά τους, ε, να συνεχίσουμε τις εργασίες και να έχουμε επαφές όπως είπε η Κομισιόν, δικαίως στην αρχή είπε σε ορισμένα σημεία η πρότασή μας μπορεί να φαίνεται επαναστατική, διότι η Κομισιόν πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η Ευρώπη, έτσι όπως έχει ε, σχεδιαστεί μέχρι στιγμή, δεν μα βοηθάει να κάνουμε βήματα προ τα μπρο. Μα βοηθάει να κάνουμε βήματα προ τα πίσω, διότι η Τελωνιακή Ένωση δεν είναι μόνο ο εξυγχρονισμό του Τελωνιακού Κώδικα. Γνωρίζουμε ότι ορισμένε από τις προτάσει μας είναι εντό εισαγωγικών μη αποδεκτές. Ωστόσο έχουμε το καθήκον να κάνουμε μια επαναστατική πρόταση, αντίδραση προς την Κομισιόν, διότι για να... πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν αλλάξει τα πράγματα δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θα έχουμε διμερεί συμβάσει σε ολόκληρο τον κόσμο, σκοτώνοντας συνεχώ την οικονομία μα. διότι δεν προστατεύουμε τα σύνορά μα. Το θέμα δεν είναι να κλείσουμε ή να ανοίξουμε εντελώ τα σύνορα. Το θέμα είναι να έχουμε κοινού κανόνε που να εφαρμόζονται και να είναι εφαρμόσιμοι και του οποίου θα χρησιμοποιήσουμε για να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία του ε, τελωνιακού κώδικα πρέπει να την αξιοποιήσουμε ώστε να καταλάβει η Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι σήμερα δεν μπορεί να αποκλείει το Κοινοβούλιο και να αφήνει στο Συμβούλιο και την Κομισιόν τα δικαιώματα να αποφασίζει ποιο θα είναι το μέλλον μας, δεδομένου ότι πόσες πολλές φορές έχουν κάνει λάθος στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κριστιανά. Εδώ ολοκληρώνεται η πρωινή μας συνεδρίαση, το πρωινό τμήμα της συνεδρίασής μας. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνος για προθεσμία, για τις τρόπολο ΓΥε 20 αυτού του μήνα στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ. Καλή όρεξη.